πλήρη σεβασμό των αρχών και στόχων της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και τώρα θα ήθελα να σας αναγγείλω ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα εξαχθεί αύριο στις 12. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το, άλλο σημείο, το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, την έκθεση της κυρία Σάιφη, εμπόριο και επενδύσεις, μοχλή ανάπτυξη της αναπτυσσόμενες χώρες. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η συγγήτρια κυρία Σάιφη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Σβέντσεν για την καλή συνεργασία που είχαμε να συμφιλιώσουμε τις, δύο, τις απόψεις των δύο επιτροπών ήταν ο κοινό μας στόχος κατά τη διάρκεια όλων των κοινοβουλευτικών μας εργασιών και θεωρώ ότι πετύχαμε αυτούς τους στόχους. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ιδιαίτερα τους σκιώδες συγητές. Ε, ε θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να είναι μια συνιστόσα της ανάπτυξης πέρα από τα παραδοσιακά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το σύστημα γενικευμένων προετοιμήσεων ή ασύμετρες εμπορικές συμφωνίες. Θα ήθελα η δική μας Επιτροπή να επιφέρει καινοτόμε προτάσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις νέες ανάγκες των εταίρων μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Για ποιο λόγο, γιατί σε αυτή την περίοδο της κρίσης κανένας προπολογισμό δεν μπορεί να επεκφύγει σοβαρών ε, περικοπών και οι γραμμές που αφορούν την ανάπτυξη πέφτουν θύμα αυτής της πολιτικής ε, λιτότητας. Γι' αυτό θα πρέπει να πειραματιστούμε με νέες μορφές ε, σύναψης εταιρικών σχέσεων όπως οι τριγωνικές εταιρικές σχέσεις, σχέσεις νότου-νότου να παράσχουμε τεχνική βοήθεια στο εμπόριο ε, ένα παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα, κατά διάρκεια μια συνεδρίαση, άκουσα έναν ειδικό εμπειρογνώμονα από τον Νότο, ο οποίο είπε ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα, αλλά εμεί δεν τα αξιοποιούμε σωστά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξελιχθούν τα κριτήρια και οι μέθοδοί μας. Αυτό είναι από τα βασικά σημεία της έκθεσής μου. Οι ίδιες οι χώρες θα πρέπει να χαράξουν κάποια στοιχεία εμπορική πολιτική. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προτείνει την ενδεδειγμένη υποστήριξη στο κατάλληλο επίπεδο, είτε σε πολυμερέ επίπεδο, στο επίπεδο του ΠΟΕ ή σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πολυμερέ επίπεδο υπάρχουν δύο προτάσεις, που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Η πρώτη αφορά την έτσι στην προσχώρηση στο, στον ΠΟΕ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. πώ μπορούν να υποφεληθούν από τι εμπορικέ αλλαγέ αν βρίσκονται στην άκρη, στο περιθώριο. Αυτή η βοήθεια δεν είναι πολύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι βοήθεια τεχνική φύσεω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να προσλάβει προσωπικό, γιατί διαθέτει ήδη εμπειρογνώμων Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, παραδείγματι και ε, κυρίως την εμπειρογνωμοσύνη στο επίπεδο των επαγματεύσεων είναι τόσο μεγάλη που θα επιτρέψει ταχύες ε, πρόοδους. Η δεύτερη είναι εξή. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει όλη τη την επιτροπή του ώστε να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες ε, τελωνιακών διευκολύνσεων και μάλιστα το ταχύτερο δυνατό. Η συνδιάσκεψη του Παλί στο τέλος αυτού του χρόνου θα μπορεί να είναι ίσως μια καλή ευκαιρία και θα ήθελα η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συμμετάσχει εκεί να ασκήσει πίεση σε περιφερειακό επίπεδο. Το κεντρικό σημείο των προτάσεών μου είναι η προώθηση της εμπορικής ολοκλήρωσης. Ένα παράδειγμα αυτό το οποίο θα, έπρεπε, θα μπορούσε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να, πάει, να ολοκληρώσει την πολιτική της είναι οι κανόνες ε, προέλευση. Όπως ήμουν εισηγήτρια της ομάδας για αυτό το κείμενο, ε, εξακολουθώ να παληθεύω σε τακτά χρονικά διαστήματα τη πρόοδου της υλοποίηση. και λυπούμε που θα πρέπει να διαπιστώσω ότι πολλές χώρες εταίροι δεν ε, το έχουν επικυρώσει και άρα λοιπόν δεν εφαρμόζεται στο σύνολο της ζώνης. Η Επιτροπή, η Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συνεργαστούν με τους εταίρους μας για να βελτιώσουν το, την εφαρμογή της προσώσης και πλήρη της αποτελεσματικότητα. Ε, ενώ βρισκόμαστε στο πλαίσιο προετοιμασίας για να ορίσουμε τους στόχους της χιλιετίας μετά το 2015, η συνεργασία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σέιφη και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους, ομι... στους στη διαδικασία ΚΑΣΔΙ. Ο κύριος ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ Θεωρώ τα σχόλια της εισηγήτριας πολύ ενδιαφέροντα και συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω πως εν ολίγης αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κινηθούμε από την βοήθεια στο εμπόριο. Ο κόσμος αλλάζει, οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, συνειδητοποιούν περισσότερο το δυναμικό τους και πρέπει να κινηθούμε από το να τους δίνουμε άμεση αναπτυξιακή βοήθεια σε κάτι που θα τους ωφελήσει στο μέλλον πρέπει να αναθεωρούμε και όλο το ζήτημα των ε, ΜΚΟ. Υπάρχουν πολλέ ΜΚΟ, όλε δουλεύουν καλά, αλλά πόσο αποτελεσματικέ είναι και πόσο είναι έτοιμε για το μέλλον. Πιστεύω πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια ε, μελέτη αξιολόγηση για τι ΜΚΟ που λειτουργούν, ίσω να τι μειώσουμε και στο μισό και να είναι πιο αποτελεσματικέ και να ανταποκρίνονται περισσότερο στι ανάγκε του μέλλοντο, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε ώστε όχι μόνο να είναι αναπτυσσόμενες, αλλά να αναπτυχθούν και όλα στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Νικολάσικ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητή Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η εμπορική και επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι άτοτε στους νόμους και στους κανονισμούς που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες. Οι στόχοι που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της Ένωσης μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμείνει στις βασικές της αξίες. Και επειδή έχει μια κάποια θέση στον κόσμο και έχει και μια ηθική ευθύνη, είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε όλες τις δυνατότητες, που, όλα τα χρήματα που υπάρχουν, ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση εν γέννη. Γι' αυτό και είμαι υπέρ αυτού του ψηφίσματος και της δουλειάς της εισηγητρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνοντα το ψήφισμα αυτό καθιστά τη θέση τη σαφή και στέλνει ένα σαφέ μήνυμα ότι θα στέκεται ότι θα στηρίζει πάντοτε τις βασικές αρχές της συνοχής και της ε, στήριξης ε, καθώς και της ε, ολοκλήρωσης των αναπτυσσόμενων χωρών στον υπόλοιπο κόσμο. Κυρία Κέλλερ. Όταν μιλάμε για το εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες πρέπει να διασφαλίζουμε ότι τα αναπτυξιακά συμφέροντα, η καταπολέμηση της φτώχειας είναι πάντως στο επίκεντρο. Ε, μας υποχρεώνει και η συνθήκη της Λισαβόνας γι' αυτό. Για να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε υποχρεωτικούς κανόνες για τις επιχειρήσεις, για την ανάληψη της κοινωνικής τους ευθύνης. Καλό την Κομισιόν την έκθεση, να ανταποκριθεί στην έκθεση της κυρίας Σαΐφη και να δει ε, με κριτικό πνεύμα την προσέγγιση των ε, συμφωνιών εταιρική σχέσης, να δει εάν εξυπηρετούν και τις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι μόνο εμάς. Μην πέσουν για μία ακόμη φορά θύματα. Χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική υπέρ της ανάπτυξης, ε, συνοχή ε, αναπτυξιακών πολιτικών. Συνοχή προς το συμφέρον της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας. Αυτό θέλουμε ως Κοινοβούλιο να εφαρμόσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Φερέιρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε οι εμπορικές οι πολιτικές και οι πολιτικές επενδύσεων στις, αναπτυξιακές, στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν πρακτικά σε επιπτώσεις τις οποίες ε, θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Ε, η περιφερειακή θέση σε, των χωρών αυτών σε σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο, η αδυναμία τους στις επενδύσεις της, ε, της που τελικά καταλήγει σε κυριαρχία των ξένων επενδυτών επιδεινώνει την κατάσταση της ανάπτυξης και επίσης επενδυνώνουν αυτές οι υποτιθέμενες ε, συμφωνίες επενδυτικές οι οποίες τελικά υποτάσσουν τις επιθυμίες τους και τις επιθυμίες των λαών τους στις, στους επενδυτές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερος χώρος για δημόσιες πολιτικές έτσι ώστε να είναι κυρίαρχες και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που, είναι στη, που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους. Είναι οι βασικές αξίες και οι δημοκρατικές οι οποίες, ε, τις οποίες αναφέρω και οποιαδήποτε πολιτική ανάπτυξη και συνεργασία αν θέλει να είναι γνήσια θα πρέπει να τις αναγνωρίσει και να τις σεβαστεί Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τελευταία μιλήτρια είναι η κυρία Μπασέσκου. Η Ένωση και τα κρατη είναι οι βασικοί δωρητές όσον αφορά την βοήθεια για το εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη διεθνού συντονισμού ε, στις ε, επενδυτικές πολιτικές των ΠΟΕ ο ΠΟΕ μάλλον θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο ως προς αυτό και συμφωνώ πως η βοήθεια για το εμπόριο που χορηγεί η Ένωση θα πρέπει να προσανατολίζεται προς χώρες που ε, το χρειάζονται περισσότερο, ιδιαίτερα οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε και αυτέ που τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε του στόχου που αναφέρονται για τη μείωση του φτώχεια, οι προσπάθειε τη Ένωση δεν αρκούν. Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη συμμετοχή όλων των άλλων περιφερειακών κρατών και η δέσμευση των χωρών BRICS για την ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Uh, και εγώ σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής για τη σημερινή μας συζήτηση είναι η Επίτροπος Κρούς. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή ε, Ανάπτυξης και την εισηγήτριά της, την κυρία Σαΐφη, για τη δουλειά που έκανε ε, για όσους δεν ήταν στην παρουσίαση της σχετικής έκθεσης ΔΕΒΑ, η Επιτροπή στην ε, εκφράζει τη λύπη του που δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση γιατί πρόκειται για μια ανακοίνωση την οποία ε, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική. Εκείνη λοιπόν που είστε μέλη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, του Διεθνού Συμπορίου θα θυμάστε ότι στην αρχή της εντολής της Κομισιόν ορισμένη δεν ήσασταν ικανοποιημένοι γιατί δίνεται δώσαμε λίγη σημασία στο εμπόριο και στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια. επιλογή αυτή όμως ήταν η θελημένη. Ο Επίτροπος Δεκούχτη θέλει να ε, ήθελε μάλλον να κάνει μια ξεχωριστή πρόταση ένα χρόνο μετά, ξεκινώντα από τη βάση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμόσει τα εμπορικά τη ε, μέσα στην παγκόσμια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή ε, συνεργαζόμαστε με χώρε που είναι πολύ μακριά είναι και είμαστε συνδεδεμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειάζεται δοθεί στην παγκόσμια αγορά η όθηση ώστε να καλυφθούν και οι ανησυχίες βιωσιμότητα. Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει νέες εμπορικές προτάσεις, συνεργαζόμαστε για να τις υποβάλουμε από κοινού μαζί με τις νέας γενιάς εμπορικές συμφωνίες. Οι περισσότερε από αυτές συνήθισαν με αναπτυσσόμενες οικονομίες και είδατε ότι οι ανησυχίες μας σχετικά με τη βιωσιμότητα ε, έχουν καλυφθεί, έχουμε δώσει προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα περιβαλλοντικά δικαιώματα χάρη στα νέα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας που σέβεται την εμπορική πολιτική. Η προτεραιότητα της Κομισιόν φέτος ε, σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι να εξασφαλίσει ότι η ένατη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ του Δεκέμβριο θα δώσει απτά αποτελέσματα προς όφελος των φτωχότερων μελών του ΠΟΕ και πιο συγκεκριμένα μέσω μιας πολυμερού συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Η απλοποίηση των ε, ε, διαδικασιών για την, το εμπόριο ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι ένας απλός και οικονομικός στόχος η μείωση των δασμών, η συμφωνία για τις ποσοστώσεις, ε, κανόνες προέλευσης κτλ. κτλ. Σε ορισμένες ε, περιπτώσεις πρέπει να γίνει αναβάθμιση για να μπορέσουν οι χώρες αυτές να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν στο παγκόσμιο αγορά. Τόσο η δική σας έκθεση όσο και η έκθεση DEVE τονίζουν την ιδιοποίηση από πλευράς της χώρας. Εμείς ε, και συνεχίζουμε να προωθούμε την ιδέα αυτή και οι ε, αποδέκτες της βοήθειας ε, θα πρέπει να μπορέσουν να εντοπίσουν τις δικές τους προτεραιότητες. Να στηρίξουμε την εμπορική πολιτική, να τη διατυπώσουμε σωστά, να δημιουργήσουμε τεχνικές ε, δυνατότητες αλλά και τεχνικές υποδομές. Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε παρά μόνο αν μας το ζητήσουν. Κάτι ακόμα θα είναι η πρόταση της Κομισιόν για μια συνολική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της της ε, υπεύθυνης ε, χρήσης των πόρων. Μια λογική και αποτελεσματική πρόταση θέλουμε να φτιάξουμε, να γνωρίζουμε ότι οι εμπορικέ ευκαιρίε αποτελούν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο και θέλουμε αυτό το δυναμικό να χρησιμοποιηθεί υπεύθυνα. Η δημόσια δαβούλευση ξεκίνησε πριν το Πάσχα και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλη του Ιουνίου. Οι απόψει του Κοινοβουλίου και των πολιτών θα εκτιμηθούν όλο ιδιαίτερος σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για το ενδιαφέρον σας για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Σας ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Κυρίες και κύριοι, η σύνοδος θα συνεχιστεί αύριο, 5η 16, 3η 16 Απριλίου 2013, από τις 9 μέχρι τις 2 και από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ. Η ατζέντα και το πρόγραμμα έχουν δημοσιευτεί.